Ε, θα κληθούμε να συζητήσουμε το θέμα της καταπολέμησης συμπορίας γυναικών και κοριτσιών για σκορπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα δώσω το λόγο στην ε, ε, συγγραφέα, η κυρία Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεκάδες ε, χιλιάδες ε, παιδιών, κοριτσιών και γυναικών ε, πέφτουν θύμα εκμετάλλευσης σεξουαλικής και εργασιακής εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι πολιτικές ομάδες αποφασίσαμε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία έτσι ώστε να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία. Ζητούμε λοιπόν σήμερα τα κράτη, από τα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν γρηγορότερα και εντονότερα έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η εμπορία. Στη Σικελία μου είπαν γιατροί, ορίστε δέστε εδώ, δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα ή ούτε ένα κορίτσι που να μην έχει ε, γίνει θύμα, πέσει θύμα βιασμού ε, στην πορεία τους ε, προς την Ευρώπη. Οι ιστορίες τους είναι συγκλονιστικές και το, μπορεί να το πει κανείς κοιτάζοντας το σώμα τους. Έφτασε η ώρα ε, να ε, ε, υλοποιηθεί, να εφαρμοστεί η οδηγία κατά, της, κατά του τράφιγγινγκ από όλες τις χώρες. Πρόκειται για μια ευρεία διαδικασία, για ένα εμπόριο το οποίο μέσα σε όρους ατιμορρησίας ε, φέρνει πάρα πολύ μεγάλα κέρδη. Πρέπει να, γίνει, να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών. Ε, να σταματήσει ε, η δυνατότητα επιγραμμικά να προωθείται αυτό το εμπόριο. Θα πρέπει να ποινικοποιηθεί και η πλευρά του αγοραστή. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι γυναίκες και τα κορίτσια αυτά να έχουν πρόσβαση σε υγεία αναπαραγωγική, συγγνώμη, σε ε, υπηρεσίες παραγωγικής, αναπαραγωγικής υγείας θα πρέπει να αισθανθούν ασφάλεια. Ε, τα όσα συμβαίνουν στην Λιβύη δεν είναι δυνατόν να τα δεχτούμε. Πρόκειται για συνθήκες ε, νέας δουλείας, πρόκειται για συνθήκες σκλαβιά και δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Σε αυτές σε αυτούς τους δρόμους της προσφυγιάς θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι εκ των συγγραφέων του κειμένου. Παρακαλώ να με αφήσετε να ολοκληρώσω, λέει κύριε Κορατσαμπίλτε. Ζητούμε νέα στρατηγική αντιτράφικινγκ ε, πέραν του 2016. Ε, και θέλουμε να συνεχίσουμε με μηδενική ανοχή. Ε, κύριε Πρόεδρε, εμείς από το 2011 προσπαθούμε να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Είμαστε εδώ και μετά το 2016, είμαστε εδώ και σήμερα το βράδυ. Τώρα πρέπει να σταματήσουμε τα λόγια και να συνεχίσουμε με πράξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Υπενθυμίζω ότι ε, είσαστε 7 εισηγητές και επομένως δύο λεπτά ο καθένας σας έχει τον λόγο έχει η κυρία Γκαρθία Πέρες για δύο λεπτά. Ινάτσε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στη σύγχρονη Ευρώπη του 21ου αιώνα υπάρχουν ακόμα σκλάβες ε, του σεξ. Υπάρχουν γυναίκες τις οποίες εκμεταλλεύονται κάποιοι σεξουαλικά αλλά και εργασιακά πάνω από 500.000 γυναίκες και κορίτσια περνάνε τα σύνορα ε, ε, ε, και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης μαφιόζικων οργανώσεων. Πρόκειται για γυναίκες οι οποίες οθούνται μέσω απειλών στην πορνεία. Γυναίκες και κορίτσια που τους κλείνουν σε οίκους ανοχής γιατί και με την απειλή ότι θα κάνουν κακό στις οικογένειές τους. Ε, κάθε μέρα εκδίδονται οι γυναίκες αυτές και τα κορίτσια αυτά σε οίκους ανοχής ε, και δεν παίρνουν τα χρήματα οι γυναίκες και οι κοπέλες αυτές. Και το τονίζω αυτό. Τα χρήματα που οι άνθρωποι αυτοί, οι πελάτες πληρώνουν στους οίκους ανοχής τελικά καταλήγουν ε, στα χέρια της και στις τσέπες της μαφίας. Νομίζω ότι εδώ είναι πολλά τα προβλήματα και επομένως εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα στην Ευρώπη για το θέμα της νομοθεσίας. Γιατί εάν δεν υπάρχουν πελάτες δεν θα γεμίζουν οι τσέπες των ε, ε καταλήλων ανθρώπων με αυτά τα βρώμικα χρήματα στη Σικελία και στην Ραγούσα πήγα τον ε, Ιούλιο και είδαμε ότι σε ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπάρχουν γυναίκες κυρίως προερχόμενες από την Ρουμανία οι οποίες δουλεύουν από τη νύχτα μέχρι την άλλη νύχτα ε, δουλεύουν 24 ώρες που λέει ο λόγος το 24ωρο και πέφτουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή και σε σεξουαλική και σε εργασιακή εκμετάλλευση ο κοινός είναι ότι πρόκειται για γυναίκες, γυναίκες ευάλωτες, γυναίκες οι οποίες έχουν ε, ε, πέσει θύματα εμπορίας. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν οι νόμοι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε όποιες δυνατότητες έχουμε. Θα πρέπει εμείς να γίνουμε η φωνή αυτών των ανθρώπων. Δεν έχουμε αυτών των γυναικών, δεν έχουμε καμία δικαιολογία πλέον να σιωπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γκέρικ για δύο λεπτά. Κύριε Γκέρκε, παρακαλώ. Κύριε Γκέρκε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τρομακτική αριθμή. Πάνω από 16.000 είναι τα ε, θύματα ε, του εμπορίου ανθρωπίνων όντων και το 1 τρίτο είναι γυναίκες. Δυστυχώς, επί της ουσίας, δεν υπάρχει τίποτα που να ε, θεωρείται αμεληταίο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλοι ό,τι είναι δυνατό ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πορνεία, την κακοποίηση των παιδιών και το παράνομο εμπόριο ανθρώπων στην Ευρώπη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταπιέζουν άλλους ανθρώπους να εργαστούν υπό ανάρμοστες συνθήκες ε, στην Ευρώπη. Λοιπόν, το να έχουμε εξαναγκαστική εργασία είναι απαράδεκτο σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, στον τομέα της καθαριότητας, στην παραγωγή κρέατος. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γίνονται θύματα εκμετάλλευσης, τους πιέζουν να δουλέψουν. Το ίδιο και στην πορνεία πάνω από το 90% των εκπονευόμενων γυναικών ε, στην Ευρώπη το κάνουν ε, παρά τη θέλησή τους. Είναι θύματα εγκληματιών. Οι γυναίκες στην Ευρώπη ε, έρχονται για να στέλνουν κάθε μήνα λεφτά στην πατρίδα τους και να ταΐζουν τα παιδιά τους με αυτή την ελπίδα. Όμως ε, εμείς ε, τις αφήνουμε να γίνονται θύματα των εγκληματιών και πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό, να είμαστε κατά της εξαναγκασμένης πορνείας και της εργασίας. Θα πρέπει να πατάξουμε το εμπόριο ανθρωπίνων όντων και να βρούμε ένα σύστημα για τα αγνοούμενα παιδιά. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι, να υπάρχει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή εμπορίου ανθρωπίνων όντων τώρα, όχι αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Μλίναρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η μεγαλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων ήταν μια τα, από τις ευχές της, για την Ευρώπη και της, για την εσωτερική αγορά. Όμως όταν βλέπουμε αυτά στις επιθυμίες να πραγματοποιούνται, ε, βλέπουμε και περιπτώσεις χιλιάδων γυναικών οι οποίες εργάζονται αναγκαστικά στον ε, τομέα της γεωργίας 12 ε, ώρες την ημέρα ε, χωρίς ε, την κατάλληλη αμοιβή. Υπάρχουν ε, εκθέσεις της αστυνομίας που μιλάνε για γυναίκες οι οποίες είναι σύγχρονες σκλάβοι. Είναι επίσημα νούμερα τα οποία μιλάνε για θύματα εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης γυναίκες οι οποίες κάποια στιγμή ε, μπορεί να μην ε, δουλεύουν γιατί είναι η ώρα να, ε, να ξεκουραστούν. Την ίδια στιγμή όμως καλούνται να γίνουν πάλι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από άλλους. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μας δείχνουν πως υπάρχει σύγχρονη δουλεία. Όχι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά σε άλλες υπήρους, εδώ μεταξύ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες οι πολίτες ε, που πλήττονται από αυτό είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά και ε, περνάνε από τα σύνορα ως θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και πρέπει τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν την ηθική επιταγή απέναντι σε αυτά τα θύματα. Να μην είναι θύματα οι άνθρωποι αυτοί της χειρότερης μορφής εκμετάλλευσης να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο, να ταυτοποιήσουμε τα ε, περιστατικά και να τιμωρήσουμε τους εγκληματίες. Ως ε, εισηγήτρια για την έκθεση αυτή θα ήθελα να μιλήσω φωναχτά για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Χρειαζόμαστε πληροφορίες για να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη τιμωρία και τις κατάλληλες επιπτώσεις ε, για τους δράστες. Ευχαριστώ και τώρα έχει το λόγο ε, η κυρία Μπιόρκ για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι εδώ και χρόνια έχουμε ζητήσει ε, μια στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών ε, αλλά δεν την έχουμε πετύχει. Τώρα έχουμε κάτι, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Ε, αυτές οι παρεμβάσεις δεν έχουν το βάρος και την σημασία και την ισχύ μιας στρατηγικής η εμπορία ε, ανθρώπων, κυρίως γυναικών και κοριτσιών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πελάτες. Είναι άνδρες ε, οι πελάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα θύματα, αγοράζουν τις υπηρεσίες αυτών των γυναικών και των κοριτσιών. Ζητούμε λοιπόν να ποινικοποιηθούν αυτού του είδους οι υπηρεσίες δηλαδή να ποινικοποιηθεί η χρήση αυτών των υπηρεσιών. Επίσης, ε, ε, από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός και το κατανοούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να αποδείξει κανείς ότι γνώριζε ή ότι δεν γνώριζε το ότι τα κορίτσια αυτά εκδίδονται μετά από ε, καταναγκασμό. Ε, θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να υπάρχει όμως μία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει παντελώς την οποιαδήποτε πώληση ε, γυναικών ή κοριτσιών ε, για ε, να απαγορεύεται η έκδοση γυναικών και η πορνεία. Θα πρέπει οπωσδήποτε και οι γυναίκες και τα κορίτσια που είναι θύματα να έχουν την δυνατότητα για ψυχολογική υποστήριξη. Κυρίως όμως και το είδαμε και από άλλες παρεμβάσεις εάν δεν μπορέσουμε να ποινικοποιήσουμε την χρήση των υπηρεσιών αυτών δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να δείξουμε θάρρος. Θα πρέπει να κλείσουμε μέσα στις φυλακές αυτούς που ε, χρησιμοποιούν την ε, την πορνεία. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Ουρτασούν. Παρακαλώ, Ερνέστο. Κοιτάξτε, η καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών ε, παίρνει διαρκώς διαστάσεις. Σύμφωνα και με τα στοιχεία ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 76% των θυμάτων ε, της εμπορίας είναι γυναίκες και κορίτσια. 16.000 περίπου έχουν φτάσει τα θύματα ε, τα τελευταία τρία χρόνια και μονάχα 3.000 είναι οι καταδίκες ε, που είχαμε μέχρι τώρα. Ξέρετε ότι ε, βεβαίω είναι πολύ μεγαλύτερα τα στοιχεία, η πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί ξέρετε ότι στις στατιστικές δεν μπαίνουν όλες οι δυνατότητες δεν μπαίνει όλη η πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση και παραβιάσεις στις γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν, ζητούν ε, άσυλο. Ξέρουμε ότι στις πολλές χιλιάδες ε, και των ε, ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ιταλίας, μέσω της Ελλάδας, είχαμε πάρα πολλά τέτοια θύματα. Επίσης ξέρουμε ότι είναι πάμπολες οι γυναίκες από την Ιγυρία οι οποίες έχουν πέσει θύματα. Επίσης ξέρουμε ότι περίπου 1560 θύματα έχουν πιστοποιηθεί ως, ε, ε, ως θύματα εμπορίας. Επίσης ε, γνωρίζομαι ότι τον Νοέμβριο είχαμε δολοφονίες ε, γυναικών ε, στην Ιταλία ε, θυμάτων δηλαδή αυτής της εμπορίας τις οποίες δολοφόνησαν οι έμποροι. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο συγκεκριμένη, να είναι πιο αυστηρή, να υποχρεώσει λοιπόν και τα κράτη-μέλη και όλους. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία ολοκληρωμένη πολιτική και όχι μονάχα κάποια μέτρα από εδώ και από εκεί. Κύριε Επίτροπε, σήμερα ε, ε, περιμένουμε να σας ακούσουμε, ε, περιμένουμε να ακούσουμε με ποιο τρόπο και με ποια μέτρα θα προσπαθήσετε να καταπολεμήσετε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, η κυρία Αγιούτο έχει το λόγο. Ντανιέλα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και σήμερα ακόμα, παρά και την οδηγία του 2011, για την ε, καταπολέμηση και τιμωρία της ε, εμπορίας ε, που ισχύει ήδη εδώ και μερικά χρόνια σε κάποια κράτη-μέλη, το φαινόμενο δεν μειώνεται. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σύμφωνα με τα στοιχεία. υπάρχει ε, ε, ε, και η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων αυτής της εμπορίας που είναι γυναίκες και κορίτσια. 76% είναι γυναίκες και παιδιά, 15% είναι ανήλικα κορίτσια ε, πρόκειται για ανθρώπους ε, που περνούν τα σύνορά μας και τελικά βρίσκονται να ζουν έναν εφιάλτη χειρότερο από αυτό που προσπάθησαν, ε, από τον οποίο προσπάθησαν να ξεφύγουν γιατί είναι θύματα σεξουαλικής ή εργασιακής εκμετάλλευσης από στοιχεία του οργανωμένου εγκλήματος. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη Τρία δις ε, ε, δολάρια κερδίζουν οι εγκληματικές οργανώσεις μόνο από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Γνωρίζομαι ότι ε, πολύ συχνά αυτή η εμπορία και η σεξουαλική και άλλη εκμετάλλευση σχετίζεται με την προσφυγιά, σχετίζεται με τα μεταναστευτικά κίνηματα που φτάνουν στις ακτές της Ιταλίας και της Ελλάδας. Δεν είναι δυνατόν όμως να αφήσουμε το πρόβλημα στους ώμους μονάχα αυτών των δύο χωρών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει αυτή η ντροπή. Είμαι υποχρεωμένη να υπενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, συγγνώμη στην Κομισιόν, ότι ε, οι εγκληματικές ε, οργανώσεις δεν αποτελούν μονάχα το σημείο στο οποίο ε, λειτουργούν οι εγκληματικές οργανώσεις. Πολλές φορές εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δημιουργούνται οι συνθήκες. Πολλές φορές αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις ψάχνουν όχι μόνο ξένες γυναίκες και κορίτσια αλλά και γυναίκες και κορίτσια εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι μονάχα ο μοναδικός ε, Εχθρό. Ε, γιατί πλέον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλέ χώρες ε, υπάρχει μια παγιοποιημένη φτώχεια η οποία σιωπηρά και σιγά σιγά διαβρώνει την κοινωνία. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή μάλιστα να σταματήσουμε την κατάσταση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε άλλο. Περιμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει ποια μέτρα θα εφαρμόσει έτσι ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα πρόβλημα αυτό. Μηδενική ανοχή όσον αφορά την εμπορία των ανθρώπων γιατί αυτή είναι μια νέα μορφή σκλαβιάς, δουλείας, η οποία κατάφορα παραβιάζει τη συνθήκη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος, εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ κύριε Αβραμόπουλο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες που ανέλαβαν αυτήν την πρωτοβουλία για την κατάθεση της προφορικής ερώτησης στην οποία πρέπει να απαντήσω. Είναι πράγματι επίκαιρη και αφορά ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και υψηλότητα στις, στα ενδιαφέροντα στις προτεραιότητες όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την διαρκή υποστήριξη που μας παρέχεται στην κοινή μας προσπάθεια να καταπολεμήσουμε αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε ότι η καταπολέμηση της, όταν προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων χρειάζονται πράξεις και όχι λόγια. Ότι οι πραγματικές πράξεις είναι αυτές που έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τις όποιες καλές προθέσεις. Έχουμε σύγχρονα σκλαβοπάζαρα. Στην Συρία, στη Λιβύη, οποιοι άνθρωποι πολλούνται και αγοράζονται σαν να είναι εμπορεύματα. Αυτό δεν θα σταματήσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι αδίστακτοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ε, αγόρια, κορίτσια, παιδιά ή ε, ευάλωτους ε, ενήλικες. Και αυτοί οι αδίστακτοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν αστρονομικά κέρδη από το, τις πράξεις τους εάν δεν τις σταματήσουμε. Τα θύματα υφίστανται βασανιστήρια, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν, απαλυνθούν και δεν μπορούν να σταματήσουν παρά μόνο να αναλάβουμε δράση τώρα. Γνωρίζετε ότι το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο τα κράτη που, βρίσκονται, που έχουν, βρίσκονται σε πόλεμο ή είναι ασταθή. Έχουμε εμπορία ανθρώπων και στην ίδια την Ευρώπη. Όπως ορθά επισημαίνει και η προφορική ερώτηση, η διάσταση του φύλου είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ιδιαίτερα ε, ξεκάθαρη στο πρόβλημα αυτό. Παρά το γεγονό ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα. Είναι επίσης γνωστό ότι η εκμετάλλευση είναι και σεξουαλική και εργασιακή. Η εκμετάλλευση την οποία υφίστανται αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι. Τι λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε. Να εστιάσουμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα εγκλήματα και να βρούμε μέτρα για την καταπολέμηση αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πράξει ή ξεκινάει, γίνεται από εδώ, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται επιτόπου, στο πεδίο, από τις αρχές, τις διοκτικές των κρατών μελών, που βεβαίως πρέπει να συνεργάζονται. Είναι λοιπόν προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτοπου στο πεδιο απο τις αρχες τι διοκτικε των κρατων μελων που βεβαίω πρεπει να διευκολύνει αυτή την επιχειρησιακή συνεργασία. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα τέτοια συνεργασία μπορούμε να το δούμε στα στατιστικά στοιχεία που μας ε, δίνει η Europol. Από το 2016 μέχρι αρχές Δεκεμβρίου του 2017 2.476 υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων παραπέμφθηκαν στη Europol. 10.664 ε, πιθανά θύματα κατεγράφησαν. Ε, στην μεγάλη τους πλειονότητα ε, υπήκο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βάση δεδομένων του Europol διαθέτει στοιχεία για περίπου 10.449 πιθανού υπέτειου αυτών των εγκλημάτων και πάλι στο, στην πλεγάλη του πλειονότητα είναι επίκοη Ευρωπαϊκής Ένωση. τελευταία χρόνια λοιπόν με την συνεργασία όλων καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ουσιαστικό, ένα ισχυρό πλαίσιο νομικό και επιχειρησιακό για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος. Τι χρειάζεται τώρα όμως. Να εφαρμοστεί στην πράξη όλο αυτό το νομικό απλοστάσιο. Αφενός και αφετέρου να αναλάβουμε δράση στοχευμένη. Προσωπικός μου στόχος και προσωπική μου δέσμευση είναι να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις. Καταπολέμηση στις διοπτικές επιχειρήσεις, καταπολέμηση αυτού του Το Προηγούμενο Δεκέμβριο παρουσίασε μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων με τα οποία θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε ε, αυτές τις εγκληματικές ομάδες, τον τρόπο λειτουργίας τους, να ενισχύσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων να βοηθήσουμε την καλύτερο συντονισμό στις προσπάθειες που γίνονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της ε, Ένωσης. Και να παράσχουμε ε, στοχευμένη οικονομική βοήθεια. Παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτού του σχεδίου και ενημερωνόμαστε και μέχρι το τέλος του 2018 θα παρουσιάσουμε και μια σχετική έκθεση στο Συμβούλιο έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον ενημερωμένα ε, στατιστικά στοιχεία τα οποία θα τα παρουσιάσουμε στην επόμενη ε, έκθεση προόδου ε, για το 2018 εστιάζοντας και ξεκαθαρίζοντας επίσης και τη διάσταση του φύλου σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ε, πολύ λεπτομεριακά πώς έχει εφαρμόσει κάθε κράτος μέλος την οδηγία για την καταπολέμηση του τράφικινγκ και εάν την έχει εφαρμόσει σωστά. Εάν διαπιστώσουμε ελλείψεις, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση. Όσον αφορά τώρα την εργασιακή διάσταση θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σύντομα την, τη δεύτερη της έκθεση για το πώς θα εφαρμόζεται η οδηγία για τις κυρώσεις στους εργοδότες που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Και προσπαθούμε να συνεργαστούμε για την, με, με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Ισότητας έτσι ώστε να μας δώσει κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις, πρακτικές συστάσεις, οι οποίες να απευθύνονται στα κράτη-μέλη για το πώς μπορούν εκεί να αλλάξουν την ομοθεσία τους και την πρακτική τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων των, των, των γυναικών, για την προστασία των, του, του, της του φύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια από το 2016 μάλλον έκανε μια συνολική επανεξέταση όλων των πολιτικών που σχετίζονται με το φύλο. Και και αυτή η εξολόγηση ε, εξέτασε όλα τα project, όλα τα έργα από το 2004 στο 2015. Ε, η μελλοντική χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντοτε θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Ε, όσον αφορά την αξιοποίηση του Ταμείου για το Άσυλο και του Ταμείου για τη Μετανάστευση, ε, έχουμε ήδη προσπαθήσει να αλλάξουμε τον τρόπο χρηματοδότηση, να φροντίσουμε χρηματοδότηση χρηματοδότηση λαμβάνει υπόψη τη πάλι τη διάσταση του φύλου. Και τέλο, ε, θα ετοιμάσουμε μια έκθεση ε, με βάση τα στοιχεία που θα μας δώσουν τα κράτη-μέλη για την περίοδο 2015-2017, συμπληρωματική. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και επίσης σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για την υποστήριξή σας. Είμαστε όλοι στην στο ίδιο στρατόπεδο, γιατί όλοι θέλουμε να σταματήσουμε αυτό το ντροπιαστικό φαινόμενο. Σας ευχαριστώ. Τώρα, ξεκινάμε την συζήτηση των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Ματέρα για 1,5 λεπτό από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε. Είναι παράδοξο που το 2018 καλούμαστε ακόμα για μία φορά να μιλάμε ε, για δουλεία. Ε, γιατί όταν μιλάμε για εμπορία γυναικών, κοριτσιών, ε, παιδιών για σκοπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης, αυτό ένα όνομα έχει, σκλαβιά, δουλεία. ναι, μιλάμε για γυναίκες οι οποίες είναι σκλάβες, ένα τέταρτο των οποίων είναι ανήλικες. 10 εκατομμύρια παιδιά εξαναγκάζονται ε, είτε να ε, εργάζονται σε συνθήκες εκμετάλλευσης ε, είτε να εκδίδονται. Σύμφωνα και με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 79% των θυμάτων της εμπορίας χρησιμοποιούνται για σκοπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να προστατευτούν τα θύματα. Ωστόσο, να μην λησμονούμε ότι αν δεν υπήρχε ε, ζήτηση δεν θα υπήρχε προσφορά. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, ε, βρούμε τρόπους έτσι ώστε να κυνηγήσουμε, να διώξουμε τους εμπόρους σε οποιαδήποτε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι διοκτικές δυνατότητες έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτό. Βρισκόμαστε στο 2018 και έχουμε ακόμα ε, ε, ε, σκλάβους και του, Η Σιμών Βέιλ έλεγε ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει παραδειγματική εφαρμογή για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να το αποδείξουμε ότι το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αρενά για 1,5 λεπτό. Μαρία, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αξιολόγηση της οδηγίας ε, για την εμπορία των ε, ε, ανθρωπίνων όντων του 2016 καταδεικνύει ότι η εκμετάλλευση γυναικών για σεξουαλικούς σκοπούς έχει τα, τα σκύπτρα ακολουθούμενη από την εργασιακή εκμετάλλευση. Στην Σικελία, στη, στον τομέα της γεωργίας, η σοσιαλιστική ομάδα έκανε μια επιτόπια έρευνα και ε, ε, αυτό το διαπιστώσαμε αλλά βεβαίως δεν είναι μονάχα στην ε, Σικελία που έχουμε τέτοιες σκλάβες και δεν είναι μόνο στον τομέα της γεωργίας και δεν είναι μονάχα Ρουμάνες είναι γυναίκες από την Ιγυρία, είναι γυναίκες και από αλλού έχουμε επίσης την εκμετάλλευση από πλευράς πολλών επιχειρήσεων οι οποίες το μόνο που θέλουν είναι να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται περισσότερο τις εργαζόμενες ή τους εργαζόμενούς τους. Ε, θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να μην μιλάμε μονάχα ε, για την σεξουαλική εκμετάλλευση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς είναι τα πράγματα στην συλλογή των μήλων ή της ντομάτας γιατί πάντα θέλουμε όλο και προϊόντα με χαμηλότερη τιμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά αυτό σημαίνει κύριε Επίτροπε ότι δουλεύουν με συνθήκες σκλαβιά οι άνθρωποι αυτοί. Επομένως εδώ έχουμε και ευθύνη και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια οδηγία αλλά τα κράτη-μέλη δεν την ε, σέβονται. επομένω. Όπω γίνεται και στις ε, κοινωνικού περιεχομένου επιθεωρήσεις να γίνονται και εργασιακές ε, επιθεωρήσεις γιατί μέσω τη προστασία των εργασιακών συνδικών θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά. Οι επιχειρήσει θα πρέπει να σέβονται του εργασιακού κανόνε. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει κυρία Φορέντσα από την ε, Γκουε. Ένα λεπτό, Ελεονόρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. εδώ ε, βρισκόμαστε σε ένα ε, φαινόμενο ε, που είναι στο σταυροδρόμι ανάμεσα από το ρατσισμό και τον φασισμό γιατί βλέπουμε ότι 76% των θυμάτων είναι γυναίκες από την Αλβανία, από την Κίνα, από την Νιγηρία και στο 80% πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Γνωρίζομαι ότι 80% των γυναικών υποχρεώνονται ε, σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτό είναι ένα στοιχείο μιας πατριαρχικής κυριαρχικής κοινωνίας ε, ε, η οποία στρέφεται κατά των γυναικών και κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ πιστεύω ότι αυτή θα πρέπει να είναι μια σε μάχη κατά του ρατσισμού και κατά του σεξισμού. Ευχαριστούμε την κυρία Ματέρα που αναφέρθηκε και στην Σιμών Βέιλ και όχι στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη συζητώντας για το θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ πολύ. Τον ε, λόγο έχει ο κύριος, ε, η κυρία μάλλον Ράιντκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε. Οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν είναι από τη φύση τους θύματα, αλλά καταλήγουν ως θύματα. Είναι ισχυρές και ανθεκτικές, πολύ συχνά όμως την χάνουν εκμετάλλευσης. Πολύ συχνά τις εκμεταλλεύεται ένα σύστημα που έχει φτιαχτεί για τους λίγους, ώστε αυτοί να βγάζουν κέρδος και για ε, να υποφέρουν οι πολλοί. Αυτό λοιπόν δεν είναι δείγμα της ε, ε, αδυναμίας αυτών των γυναικών, οι οποίες την χάνουν εκμετάλλευσης. Είναι δείγμα της δικής μας αδυναμίας που αφήνουμε τόσες γυναίκες και παιδιά να μην ζουν ελεύθερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη λοιπόν πρέπει να πάει από τη μια πλευρά στην άλλη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ αδύναμα γιατί δεν μπορούν να εφαρμόσουν μια οδηγία η οποία πρέπει να εφαρμοστεί και η Κομισιόν πρέπει να γίνει πιο ισχυρή. Πρέπει να ενισχύσουμε τα σύνορα, πρέπει οι δράστες να τιμωρούνται, πρέπει να εκπαιδεύσουμε καλύτερα την αστυνομία και το δικαστικό προσωπικό για να αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις εμπορίου ανθρωπίνων όντων. Και είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουμε τα θύματα που πολύ συχνά μένουν μόνα τους. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι η δουλειά που δεν έχουμε τελειώσει για τον αιώνα αυτό. Ας τα διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα και ας φτιάξουμε ένα σύστημα ανθεκτικό. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Νογμανό εκ μέρου ε, της Ομάδας για της Ευρώπης, ε, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως ε, το είπε και η Κομισιόν ε, τα 15.000 θύματα του εμπορίου ανθρωπίνου όντων ε, στην, ε, στο έτος 2013-2014 ήρθαν εκτός Ευρώπης. Το γεγονός που λέει και η ίδια η Κομισιόν ότι τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων εκμεταλλεύονται την προσφυγιά και την παράνομη μετανάστευση, τους πιο ασθενείς, τις γυναίκες και τα παιδιά. Ε, είναι ε, εμφανές, βλέπουμε ότι εκμεταλλεύονται επίσης το σύστημα ασύλου. Ε, έτσι, στην απάντηση του Ιουλίου του 2017 η Κομισιόν στρέφεται κατά των κρατών μελών και λέει ότι δεν εφαρμόζουν σωστά την σχετική οδηγία. Δεν μπορούμε παρακαλώ, παρακαλώ παρά μόνο να μιλήσουμε για την πλήρη απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχουμε μια ανευθυνότητα ως προς την μεταναστευτική πολιτική, έχουμε αυτή τη μοντέρνα δουλεία και την σεξουαλική εκμετάλλευση που αγγίζει κυρίως παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο λόγος στην κυρία Τροζίσκη εκ μέρου ε, της ομάδας της Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε το εμπόριο ανθρωπίνων όντων, η πορνεία, η εξαναγκαστική εργασία είναι μια πραγματικότητα σε όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο. Όπως είπαν και προηγούμενοι, είναι το ίδιο παρούσε με την εμπόριο ναρκωτικών. Ε, ε, βλέπουμε κάθε μέρα γυναίκες και παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα να γίνονται θύματα εκμετάλλευσης. Ε, το 65% είναι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι άλλες από μακρινές χώρες. Η UNICEF μιλά για τις γυναίκες από την Ιγυρία. Τι προτείνετε εσείς. Ε, ζητάμε η Κομισιόν να δώσει περισσότερες κυρώσεις στα κράτη-μέλη που δεν ε, σέβονται τη στάδια και δίνα ε, οδηγίες, σαν αυτό να βοηθούσε τα θύματα. Και πραγματικά... Δεν μιλάτε για τη Σέγγεν, για το γεγονός ότι υπάρχει μια βοήθεια προς τους διακινητές. Η Κομισιόν αύξησε τις ποσοστώσεις των μεταναστών να έτσι ώστε ε, να τους ε, βοηθήσει να γίνουν και σκλάβοι και ε, θύματα πορνείας. Πραγματικά πρέπει να ρυθμίσετε μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να είχε ως τώρα ρυθμιστεί χωρίς άλλο πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Ντότς εκ μέρου των μη εγγεγραμμένων για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σοβαρό έγκλημα το οποίο μπορεί να διαπραχθεί εναντίον ενό ανθρώπου οποιοδήποτε υπηκότητα ή ηλικία. Είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμω το 70% των θυμάτων εκτιμάται ότι παγκοσμίω είναι γυναίκε και κορίτσια. Τα στοιχεία για το έγκλημα μας δείχνουν ότι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες θύματα. ήταν μόνο η κορυφή του παρογούβανου. Τα προηγούμενα στατιστικά στοιχεία που μα μιλούσαν μόνο για 10-13.000 θύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόσφατα εγκρίθηκε μια νέα νομοθεσία στην ε, Ιρλανδία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα, Βόρεια Ιρλανδία, η οποία μα δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τα θύματα. Με, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποζημίωση των θυμάτων, την υποστήριξή του, τη δυνατότητα να ε, δοθούν κάποιοι, η δυνατότητα και δαιμόνων για τα παιδιά, ή επίση διευκολύνσεις όσον αφορά την κατάθεση των, τις του τους καταθέσεις. Είναι μεγάλη πιθανότητα να, βρει να συναντήσει κανείς ένα θύμα του τράφικινγκ. Ο μόνο τρόπο στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα αυτό είναι η καλύτερη εκπαίδευση. ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σουηδρόβα για ένα μισή λεπτό. Ε, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ λυπηρό ε, όταν ακούω σήμερα εδώ ότι δεν είναι λίγα τα θύματα του εμπορίου ανθρωπίνων όντων. Οι στατιστικές που μιλάνε μέχρι και για δύο εκατομμύρια είναι πολύ λυπηροί διότι στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι αυτοί είναι παιδιά και γυναίκες. Υπάρχουν λοιπόν ε, διάφοροι κλάδοι όπως η γεωργία ή η οικιακή βοηθή ε, όπου οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία. Αν το δούμε και γεωγραφικά η Αλβανία, η Κίνα, το Μαρόκο, η Νιγηρία και το Βιετνάμ είναι οι χώρες προέλευσης αυτών των γυναικών. Αυτά τα θύματα ανθρωπίνου ε, εμπορίου ε, είναι πραγματικά κάτι που δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε. Πρέπει να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις. Η δημοκρατία της Τσεχίας αποτελεί και στόχο αλλά και χώρα διαμετακόμισης. Δεν είναι χώρα προέλευσης μόνο. Ε, χρειαζόμαστε προστασία και βοήθεια για τα θύματα, να έχουμε ειδικά προγράμματα και έχουμε και καλή συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με μη κερδοσκοπικέ οργανώσεις, οι οποίες είναι ένα σημαντικός εταίρο μας ε, στην πάνταξη αυτή της μορφή εμπορίου. Γι' αυτό λοιπόν ε, προτείνω και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν πιο στενά με τις μη ε, κερδοσκοπικές οργανώσεις γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλές δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο που θα πρέπει να ενισχυθούν για να έχουμε πιο απτά αποτελέσματα. Να μπορέσουμε να ορίσουμε πιο απτά το πεδίο. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο στον κύριο Μαρτάν για ένα μισή λεπτό. Παρακαλώ, Εντουάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι αξίες μας έχουν κάποιο κόστος, έχουν κάποια τιμή. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχουν καθορίσει κάποιοι αυτή την τιμή. Είναι, το κιλό ε, μιας, ε, είναι η τιμή ενός κιλού ε, μικρών ντομάτων στο, από την Σικελία. Αυτές, αυτά τα ντοματίνια λοιπόν είναι αυτά τα οποία είναι το αποτέλεσμα μιας κοινωνικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών από την Ιγερία, την Τινησία και την Ρουμανία που όπως υπόθηκε και προηγουμένως οργανώνεται η εκμετάλλευση αυτή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ε, ε, πολλές φορές. Εμείς ε, συναντήσαμε γυναίκες οι οποίες ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον αλλά δεν μπορούν να το έχουν αυτό το καλύτερο μέλλον. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να κατεδικαστούν αλλά και οι καλές προθέσεις και τα καλά αισθήματα βέβαια δεν μπορούν να σταματήσουν την σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση. Σας ζητώ λοιπόν κύριε Τρόπε να μας παρουσιάσετε την στρατηγική σα ε, για την καταπολέμηση τη εμπορία γυναικών και κοριτσιών που διαρκώ εξαπλούται και αυξάνεται. Είναι πλέον ε, η κατεπίγουσα η κατάσταση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστούν κυρώσει οι χώρε οι οποίε δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε και εμεί όλοι να έχουμε περισσότερα μέσα για να καταπολεμήσουμε την πληγή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κούνεβα. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ κυρία Κούνεβα κύριε επίτροπε υπάρχουν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στα θερμοκήπια της ιταλίας και στα χωράφια μανιταριών της ολλανδίας κακοποίηση εργαζομένων στις καλλιέργειες σπαραγγιών της τσεχίας και τις καλλιέργειες φράουλας της ελλάδας πριν μερικά χρόνια. το τράφικινγκ και η εργασιακή εκμετάλλευση ντροπιάζουν την ευρώπη δεν τροφοδοτούν μόνο τη βιομηχανία του σεξ αλλά και τη γεωργία την κτηνοτροφία τις κατασκευές τον τουρισμό την παροχή φροντίδας. η ευρώπη δεν μπορεί να είναι περήφανη με την ανάπτυξη που συνδέεται με αυτό το σύγχρονο δολεμπόριο. η επιτροπή ελέγχει αν εφαρμόζονται οι οδηγίε σε την εμπόρια ανθρώπων και του εποχιακού εργάτες ή ενδιαφέρεται μόνο για του δημοσιονομικού κανόνες. Επειδή το πρόβλημα πρέπει να λυθεί, χρειαζόμαστε έξυπνους ελέγχου εργασία, όπω τόνισα και στην έκθεσή μου για το οικικό προσωπικό, νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες για την εργασία των μεταναστών, και το πιο σημαντικό διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων για να μπορούμε να μπούμε και πραγματικά στο 21ο αιώνα. Μόνο έτσι μπορεί να σπάσει ο φόβος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. And now I give ε, θα δώσω κυρία για δύο λεπτά. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Πάρκη για δύο λεπτάκια. Ευχαριστώ. Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση έχει αυξηθεί. Το 2016 εκτιμάται ότι το ένα από τα, στα ε, θύματα ήταν παιδιά. Όμως γνωρίζουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι μικρότερα από το πραγματικό πρόβλημα, γιατί βασίζονται μόνο στις καταγγελίες. πολλές, ε, και, και εκτός αυτού υπάρχουν πολλές συχνά ε, αναντιστοιχίες, ε, λάθη. Πρόκειται για μια νέα μορφή δουλεμπορίου. 10.000 παιδιά κατά τη διάρκεια του 2015, σύμφωνα με την Europol, εξαφανίστηκαν στην ε, Ευρώπη. Κατά πάσα πιθανότητα αυτά οδηγήθηκαν είτε σε εξακαναγκαστικούς γάμους είτε σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι ιδιαίτερα ευάλωτοι ε, ε, πληθυσμοί των προσφύγων και των μεταναστών είναι εκείνοι οι οποίοι πέφτουν θύματα. Έχουμε εγκληματικές ομάδες οι οποίες εκμεταλλεύονται τη δυνατότητά τους να, περνούν τα σύνορα εύκολα και στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν τους ανθρώπους αυτούς σαν πιόνια στο, ε, στο, στο, στο οργανωμένο έγκλημα, στις μαφιόζικες πρακτικές, γιατί για αυτούς δεν είναι τίποτα, είναι απλώς αναλώσιμοι. Πρέπει να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στην πραγματικότητα διευκολύνει τους εγκληματίες. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν δίνεται η δυνατότητα στις διοικητικές αρχές των κρατών μελών να κάνουν ελέγχους και άρα δεν πρέπει να μα παραξενεύει το γεγονό ότι οι κλιματικέ ομάδε αυτό το εκμεταλλεύονται. Δεν είναι εύκολο το θέμα. Κάθε φορά που κάνουμε, τη συζήτηση, κάθε φορά κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή την ουσία του προβλήματο και δεν καταλήγουμε σε αποτελεσματική δράση. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χέντ για δύο λεπτά. Παρακαλώ, κυρία Χέντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν ε, έχει πάρει εν τέλει μέτρα ε, για να αντιμετωπίσει το θέμα της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών. Επανειλημμένο ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος μας έχει υποσχεθεί ότι θα πάρει μέτρα, αλλά παρόλα αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμα τα μέλη αυτά. Δεν έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Δεν βλέπουμε δηλαδή μία στρατηγική από πλευρά της Κομισιόν η οποία να μπορεί ε, να αλλάξει την κατάσταση. Εδώ και δέκα χρόνια συζητούμε το θέμα της ε, εμπορίας ε, ανθρώπων στο Κοινοβούλιο και διαρκώς υπάρχουν άνθρωποι και περιστάσεις οι οποίες μας σταματούν. Έχουμε προσκόμματα διαρκώς ενώ αυτό το θέμα της εμπορίας είναι ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει τα στενά εθνικά σύνορα. Είναι ένα υπερεθνικό πρόβλημα άρα χρήζει υπερεθνικής λύσεως γιατί πραγματικά με την στάση μας ε, είναι σαν να δίνουμε, την, ε, σαν να λέμε στους ε, εγκληματίες και τους κακοποιούς συνεχίστε, θα συνεχίσετε ανενόχλητοι, κανείς δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει. Όχι, θα πρέπει οπωσδήποτε να σκύψουμε πάνω στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και επομένως αυτό σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την ζήτηση, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε βοηθήσουμε τα χρήματα θα πρέπει ε, να στραφούμε εναντίον αυτών των κακοποιών και των εγκληματικών οργανώσεων ε, θα πρέπει να στηρίξουμε τις, ε, τα θύματα και κατά την διάρκεια αλλά και των ερευνών αλλά και των δικαστικών διεργασιών αλλά και μετά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διοκτικών και δικαστικών αρχών κτλ. Δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε άλλο στην Ευρώπη αυτό το εμπόριο. Πότε επιτέλους η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια πραγματική στρατηγική για πραγματική καταπολέμηση της εμπορίας. Αναρωτιόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Για ένα λεπτό, Ζωάο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε η σεξουαλική εκμετάλλευση και το οργανωμένο έγκλημα γύρω από αυτήν έχει μεγαλύτερα κέρδη ακόμα και το εμπόριο, από το εμπόριο ναρκωτικών. Χρησιμοποιούν επίσης τους φορολογικούς παραδείσους για να ξεπλένουν τα κέρδη από το εμπόριο αυτό. Και ε, ε, το, το, το πρόβλημα είναι ευρύτατο. Υπάρχουν, ε, υπάρχει η πορνεία, υπάρχει η εκμετάλλευση των ανθρώπων στις εργασιακές, στις στο εργασιακό επίπεδο, υπάρχουν εξαναγκαστικοί γάμοι. Ε, έχει λοιπόν πολλές μορφές η εκμετάλλευση. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η πορνεία μπορεί να είναι εθελούσια ή να είναι ε, δικαίωμα, μια, η επιλογή μιας γυναίκας. Ε, εμείς διαφωνούμε, εμείς πιστεύουμε ότι πρόκειται πάντοτε για, για μια εκμετάλλευση των πλέον φτωχών γυναικών, των πλέον ευάλωτων γυναικών. Είναι πάντοτε μια παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επομένως θα πρέπει να αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, όπως ορισμένες από αυτές που ε, γίνονται αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία για να νομιμοποιηθεί η πορνεία. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Παντσέρη για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε όπως ε, υπόθηκε ήδη, δεν ε, ε, χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ μακριά για να βρει, να βρει ιστορίες σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης. Καθημερινές είναι αυτές οι ιστορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θύματα πλήθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις δε είναι γυναίκες, κορίτσια και παιδιά. Για τα περισσότερα από τα θύματα αυτά, ε, η εκμετάλλευση δεν είναι μόνο εξωσεξουαλική αλλά και εργασιακή. Χείριστε σε συνθήκες εργασίας, ατελείωτες ώρες εργασίας ε, και τη μισθή είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ε, με απάνθρωπες συνθήκες στην γεωργία. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα πέθαναν ε, οι εργαζόμενοι. Συνέβη αυτό ε, το 2015 στην Απουλία. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος 29 ετών γιατί έκανε συγκομιδή στον τρίγο και ενώ ήταν νέος άνθρωπος ε, λόγω των εξουθενωτικών συνθήκων έχασε τη ζωή του. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ε, και την πλευρά όλων αυτών των επιχειρήσεων που είναι συνένοχες. Είτε πρόκειται για μεμονωμένε επιχειρήσει, είτε πρόκειται για επιχειρήσει που ανήκουν σε εγκληματικά δίκτυα. Χρειαζόμαστε επίση πολιτικές κατάρτισης οι οποίε θα δίνουν μεγαλύτερε δυνατότητε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν κοινωνικές πολιτικές. Ε, χρειάζονται ε, πολιτικές ε, πιο υποχρεωτικές και δεσμευτικές. Τέλος, κύριε, Πρόεδρε, Επίτροπε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τα λόγια και να περάσουμε στις πράξεις. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Βαγίνα για ένα λεπτό. Άγχελα Βαγίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η εργασιακή εκμετάλλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς είναι ε, καθημερινό ε, φαινόμενο και η Υπηρεσία ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται σε αυτό και μάλιστα και στην κινητικότητα την εργασιακή η οποία τελικά υποθάλπτει την εργασιακή εκμετάλλευση. Δεν είναι σωστές οι συνθήκες εργασίας και ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι ισχύουν ε, οι νόμοι η εκμετάλλευση υπάρχει και αυτή η εκμετάλλευση έχει τις περισσότερες φορές γυναικείο πρόσωπο 76% ε, δηλαδή 4 στα 5 θύματα ε, είναι γυναίκες ή κορίτσια. Επομένως χρειαζόμαστε όχι απλώς δηλώσεις προθέσεων αλλά συγκεκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένες πολιτικές καταπολέμησης της εμπορίας των ανθρωπίνων όντων. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο διάλογο, χρειαζόμαστε παρακολούθηση των καταστάσεων από κοντά. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Ward για 1,5 λεπτό. Τζούλη παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αύξηση του εμπορίου ανθρωπίνων όντων είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ανισχύει ιδιαίτερα εμάς τους, ε, τις φεμινίστριες ειδικά διότι γυναίκες είναι αυτές που την χάνουν να γίνονται θύματα αυτού του εμπορίου, κυρίως για σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτό αντιφάσκει πλήρως ε, με τις αξίες μας, όπως και με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Πολλές φορές ακόμα λοιπόν θα δούμε γυναίκες ε, να μην ε, έχουν τη δυνατότητα να είναι άνθρωποι. Να υπογραμμίσουμε την κατάσταση των εργαζομένων στη σεξουαλική ε, βιομηχανία. Οι περισσότεροι φόνοι ας πούμε γίνονται κατά των γυναικών οι οποίοι είναι ήδη θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα βήματα που έχει κάνει η Κομισιόν για να ολοκληρώσει και να τελειώ, δώσει ένα τέλος σε αυτό το εμπόριο. Πραγματικά είναι κρίμα να ε, Προσποιήστε ότι παίρνετε σοβαρά το θέμα όταν έχουμε τόσους μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη και πραγματικά όταν έχουμε ένα τόσο ε, σοβαρό ζήτημα, ειδικά για τις γυναίκες και τα παιδιά. Περιμένω τις απαντήσεις σας, Επίτροπε. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο η κυρία Μπόιλεν για ένα λεπτό. Παρακαλώ, Λίνα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Το 2018 έφτασε ήδη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ακόμα, ε, υπάρχουν ακόμα σεξουαλική εκμετάλλευση είναι σκλάβοι και ε, οι γυναίκες και τα παιδιά είναι η πλειοψηφία αυτών. Ε, όπως είπαν και προηγούμενοι, ε, σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να ξεχνάμε τις γυναίκες και τα κορίτσια που είναι ευάλωτες και δεν είναι αποδεκτό να αυξάνεται η εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών και σε εργασιακό επίπεδο. Είναι απαραίτητο και απιτακτικό να λάβει δράση η Ευρώπη. Οι δράστες πρέπει να τεθούν πρώτων ευθυνών τους, να τους φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης και να ποινικοποιηθούν οι εταιρείε αυτές που χρησιμοποιούν ε, την εργασία ε, με τρόπο τέτοιο και το ανθρώπινο εμπόριο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα τις αντίστοιχες οδηγίε για τους εποχιακούς εργαζόμενους, ε, για το εμπόριο ανθρωπίνων όντων έτσι ώστε να μειώσουμε το εύρος της βλάβης και να πατάξουμε την ανθρώπινη δουλεία για πάντα. Ευχαριστώ και τώρα ανοίγω τη διαδικασία του ΚΑΤΣΛΙΑΗ. Έχω λάβει πέντε αιτήματα σχετικά και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζαμπόρσκα. Για ένα λεπτό παρακαλώ κυρία Ζαμπόρσκα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πριν από 13 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρευρέθησε μια αντίστοιχη συζήτηση με τη σημερινή και δυστυχώς συνάδελφοι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ακούσαμε πάλι τα ίδια ότι είναι κατά κύριο λόγο γυναίκε στα θύματα. Γνωρίζουμε ότι από πέντε ανατολικέ ευρωπαϊκέ χώρε, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και άλλε, ε, προέρχονται κυρίω τα θύματα. Είναι δηλαδή αυτέ που ονομάζουμε οι νέε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εμπορία ανθρώπων ανθεί όταν υπάρχει φτώχεια, όταν υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ανισότητες. Και όσο συνεχίζουν αυτές οι τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, θα, όσο συνεχίζουμε να έχουμε δύο Ευρώπες στην πραγματικότητα, δεν θα αλλάξει το πρόβλημα. Η πραγματική ενότητα δεν έρχεται μόνο με το να κρεμίζουμε τους, τους, τα τείχη. Χρειάζεται πραγματική αλληλεγγύη. Χρειάζεται πραγματικός σεβασμός της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου και συνεργασία πέρα και πλέον πέρα από τα σύνορα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον, ε, στην Κατερίνα Κινήση. παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η εμπορία γυναικών ε, και κοριτσιών, γιατί αυτά είναι τα περισσότερα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντί να μειώνεται και παρά ε, την οδηγία του 2011 παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση ε, οπωσδήποτε και λόγω της προσφυγικής κρίσης στα πλαίσια της οποίας έχει αυξηθεί με ιδιαίτερο τρόπο ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ε, στις Σε πολλές ε, περιπτώσεις και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται αυτά τα ανήλικα παιδιά ε, πέφτουν στα δίχτυα και στα νύχια διαφόρων εμπόρων που τα εκμεταλλεύονται σεξουαλικά και εργασιακά. Θα πρέπει οπωσδήποτε όλες οι χώρες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και σωστά την οδηγία. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν οι διαδικασίες των θυμάτων καθώς επίσης και οι διαδικασίες επιμέλειας και κυδαιμονίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Μαριάς ε, για ένα λεπτό παρακαλώ Νότι. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών για σκοπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι πρέπει να ληφθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα διαπιστώθηκε ότι το 76% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν γυναίκες ενώ το 15% παιδιά. προέρχονται από τη ρουμανία τη βουλγαρία τις κάτω χώρες την ουγγαρία και την πολωνία. είναι δεδομένο ότι αυτή η εκμετάλλευση ιδίως η εργασιακή εκμετάλλευση επικεντρώνεται στον γεωργικό τομέα. θα πρέπει λοιπόν τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2011/36 να τιμωρηθούν οι δουλέμποροι και να υπάρξει δίωξη των σωματεμπόρων. ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξουν και συνεργασίες των κρατών για να αντιμετωπίσουν αυτή την διασυνοριακή εμπορία ανθρώπων. ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Μπιλμπάο Μπαραντίκα, για ένα λεπτό. Η Τσασκούν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το πρόβλημα, κύριε Επίτροπε, ε, στην ουσία συνδυάζει οργανωμένα ε, διεθνή δίκτυα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης ε, ανταπόκρισης σε τοπικό και περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και προσέγγιση από πλευράς υγειονομικής και κοινωνικής. Χρειάζεται επομένως πολύ καλή προετοιμασία της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση αυτής της πληγής ε, θα πρέπει να ε, προβλέπονται επομένως και συγκεκριμένα μέρη. Αυτό ε, το άλλωστε το τέταρτο τετραετές πρόγραμμα για την προστασία των εποχικών εργαζομένων ας πούμε στη χώρα των Βάσκων με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένα λόγια. Επίσης θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των εξαφανισμένων ε, ασυνόδευτων ανηλίκων ε, γιατί ξέρουμε ότι, ε, παίζει ρόλο και όσον αφορά τις παράνομες υιοθεσίε και όσον αφορά την παράνομη διακίνηση οργάνων. Ο κύριος Επιτίδιος για ένα λεπτό. Γιώργο παρακαλώ. Η εκμετάλλευση ανθρώπων και κυρίως γυναικών και κοριτσιών για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία έχει τις ρίζες στην αρχαιότητα αλλά δυστυχώς στη σημερινή εποχή έχει λάβει την μορφή μιας επικερδούς οικονομικής επιχειρήσεως. η κατάσταση αυτή αποτελεί στίγμα για τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μας. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη αλλά και άλλες χώρες να λάβει δραστικά μέτρα ούτως ώστε αυτή η απαράδεκτη κατάσταση αρχικώς να μεν περιοριστεί στο τέλος δε να εξαλειφθεί δεν αρκεί να αναφέρεται η ευρωπαϊκή ένωση και να επικαλείται τα άρθρα 5 και 31 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η δουλεία και η καταναγκαστική εργασία και αναγνωρίζεται στον εργαζόμενο το δικαίωμα για δίκαιη προσφορά και συνθήκες εργασίας. Πρέπει να εφαρμόσει αυστηρούς ελέγχους στις χώρες εκείνες στις οποίες είναι δεδομένες τόσο η σεξουαλική όσο και η εργασιακή εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών και παράλληλα να εμποδίσει την ανεξέλεγκτη δράση των δουλεμπόρων και των σωματεμπόρων. τέλο πρέπει να θεσπίσει αυστηρού νόμου οι οποίοι θα προβλέπουν εξοντωτικέ ποινέ για αυτού του εκμεταλλευτέ που είναι αδίστακτοι και απαράδεκτοι. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Αβραμόπουλος εξ ονόματος της Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για άλλη μία φορά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ουσιαστική και χρήσιμη συνεισφορά σας. Μα χαρά μου άκουσα και δεν το κρύβω ότι όλοι εδώ στην αίθουσα συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Αυτές που εγώ εξέθεσα με την εισαγωγική μου ομιλία. Έχουμε μια ξεκάθαρη στάση βασισμένη στην αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να δράσουμε. Με την πάροδο των ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν επιδείξει μια μεγάλη δέσμευση να πατάξουν τους αδίστακτους εγκληματίες να προλαμβάνουν το έγκλημα και το πιο σημαντικό να προστατεύουν τα θύματα. Έχουμε εξελίξει μια ισχυρή νομοθεσία και πολιτικές. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη μόρφωση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνουμε και πιο επιχειρησιακοί στο έργο μας. Μόνο αν όλοι εργαστούμε μαζί, οι Προεδρία του Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κοινωνία των πολιτών και οι οργανισμοί μας, δηλαδή, μόνο τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά στο πεδίο και είμαστε αποφασισμένοι να το πράξουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν είναι αφοσιωμένη στην ε, αναβίωση των προσπαθειών. Θέλουμε να θέσουμε δράσεις προτεραιότητας οι οποίες ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Εγώ προσωπικά, όπως το είπα και το υπογράμμισα και στην αρχή, είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα το πετύχουμε και, είμαι και δεσμεύομαι προς αυτό στα τέλη του έτους, σίγουρα, ε, αργότερα μάλλον μέσα στην πάροδο του θα ενημερώσω το Κοινοβούλιο για όσα έχουμε επιτύχει. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.